εργασίας ε, θα οδηγήσει στην υπερψήφιση των εκθέσεων και θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τη συνεργασία τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ζουαντό. Για τέσσερα λεπτά ο κύριος Δεζίρ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πίτροπε,